we have a Uh, so good afternoon, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ που ήσασταν στην ώρα σας. Με συγχωρείτε που ξεκινάμε καθυστερημένα. Σας παρακαλώ μπορείτε να ε, κάνετε λίγη ησυχία. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για το 2012. Έχουμε άλλες τρεις ψηφοφορίες πριν τις διακοπές. Νομίζω ότι εργαστήκαμε πολύ σκληρά όλοι. Αρχίσαμε με κάποια καθυστέρηση. Είναι γιατί υπήρξε μια απρόοπτη εξέλιξη όσον αφορά το θέμα του κυρίου Μπαλντασάρε για την Τελωνιακή Ένωση. Θα σας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Υποβάλαμε μία πρόταση τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις πληροφορίες σήμερα, αλλά θα αφήσω τον κύριο Μπαλντασάρε να σας εξηγήσει τι πρόβλημα έχουμε και να σας κάνει μια πρόταση που ελπίζω να δεχτείτε. Ο κύριος Μπαλντασάρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πριν από την ε, διέρεση του προγράμματος Φίσκους υπήρχε αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Μετά την, ε, το διαχωρισμό των δύο προγραμμάτων ξεκινήσαμε χωρίς γνωμοδότηση. Ωστόσο η συγκεκριμένη Επιτροπή εξέδωσε μια γνωμοδότηση την οποία μας την έδωσε υπήρχε ένα κομμάτι που αφορούσε το φίσκους τα φορολογικά, αλλά ε, υπήρχαν και τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμού, πάνω στις οποίες έγινε επίσης ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία δεν έχει πια σημασία, δεν έχει πια κάποια αξία. Ε, είναι μια γνωμοδότηση για το σύνολο του προγράμματος. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα χωρίστηκε στα δύο. Όπως και να έχει, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα, ενημερώθηκα από την γραμματεία πριν από λίγο γι' αυτό. Ε, εν αναμονή της λύσης του προβλήματος κάνω μια πολύ απλή πρόταση. Ας ψηφίσουμε εμείς όλη την έκθεση. Ας αποφύγουμε να ψηφίσουμε την τελική πρόταση ώσπου να ξεκαθαριστεί εάν αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι έγκυρη ή όχι. Αν είναι έγκυρη πρέπει να δούμε τις τροπολογίες της Επιτροπής και να ψηφίσουμε μετά επί του συνόλου. Εάν δεν είναι έγκυρη, τότε τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε επί της έκθεσης χωρίς τη γνωμοδότηση και έτσι θα λυθεί αυτό το ακαθόδε ζήτημα. Ευχαριστώ. Νομίζω πως είναι πολύ λογική πρόταση. Συμφωνείτε, οι συντονιστές μήπως έχουν καμία άλλη άποψη, ωραία. Να προχωρήσουμε με αυτή τη βάση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον η Επιτροπή Προϋπολογισμών καταφέρνει να καταφέρνει να ε, είναι στο ίδιο μήκος κύματο με εμά. Λοιπόν, είναι κανείς από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κυρία Πέντεργας, νομίζω ότι θέλετε να παίξετε ρόλο διαμεσολαβητή. Είναι κανείς άλλος από εμάς εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κανείς δεν το παραδέχεται. Ωραία. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Μπαλτασάρε. Έχουμε πρώτα απ' όλα την τροπολογία 44. Φάντε Κάμον, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 46, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική α που βλέπετε υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 17 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 κομφεράτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 του εισηγητή και 6 του κ. κοφεράτη, υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται 70 κοφεράτη υπέρ κατά αποχές 19 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ Α, με συγχωρείτε. Τροπολογία 21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71. θέλει να πει να βάλουμε ως ε, συμπλήρωση τη λέξη ενδεικτικό. Ενδεικτικό λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχή. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Υπέρ. θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για να ζεσταθούν τα δάχτυλά σας. 73 λοιπόν. 24, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, προτρέχω. 24 λοιπόν, του εισηγητή. Πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 72, κοφεράτη. Άρχεται για την 72. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται. Ανθρωπολογία 25 του Σίγητη υπέρ. Μου συγχωρείτε, χρειάζομαι διακοπές. 73. Κοφεράτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 του συγητή είμαι σε δηλογικές σκέψεις υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 2 ε, του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 είναι συμβατή με τη 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 Βαντερκάμεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 συμβατή με την 3 υπέρ κατά αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι μόνο αν συμφωνούν οι υπόλοιποι Ωραία. Λοιπόν, η πρόταση είναι να τις ψηφίσουμε από κοινού, αλλά τώρα περνάμε στην τροπολογία Σμιτ. Ψηφίσαμε 38. Το θέμα ήταν ε, να περάσουμε για όλη τη σελίδα. Αλλά θα είχαμε τελειώσει τώρα. Όλοι έχετε συν μέχρι και την 11. Όχι, όχι, η 9 για μένα δεν είναι έτσι. Ας συνεχίσουμε όμως έτσι. Θα είχαμε φτάσει τώρα. 39 Σμιτ. Συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4, 4 του συγκεκριτή υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 κοφεράτη υπέρ Α, υπάρχουν ορισμένοι κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 αποσύρεται 33 του συγκριτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία. Ολοκληρώσαμε αυτή την ψηφοφορία και μόλις ο κύριος Μπαλτασάρε καταλήξει τις διαπραγματεύσεις του Μητροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να ξανακάνουμε μια σύντομη ψηφοφορία για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Οπωσδήποτε όμως σα αξίζει ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας επ' αυτού. Ωραία. Ωραία. Καλή προθέρμανση. Τώρα να ψηφίσουμε για τον ενιαίο φορολογικό κώδικα. Τελωνιακό συγγνώμη κόρηκα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, παρακαλώ έχετε το λόγο για να ε, εισαγάγετε, να μας παρουσιάσετε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους συγητές και τους κοιόδης ε, με τους οποίους ε, συνεργαστήκαμε πολύ θετικά, δημιουργήσαμε κλίμα πλήρους εμπιστοσύνης. συνεργασίας και διαφάνειας. Ελπίζω αυτή η ατμόσφαιρα να συνεχίσει να υφίσταται και κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας, τη Γραμματεία της Επιτροπής, όλους μας τους βοηθούς και καταλήγοντας για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για το λευκό λεγόμενο τμήμα του κειμένου όπως επανειλημμένα είπαμε, είμαστε στην διαδικασία αναδημιουργίας του κειμένου και υπάρχει μια διάκριση για τον τρόπο υποβολής τροπολογιών ανάλογα με το εάν είμαστε στο γκρι τμήμα του κειμένου που εύκολα μπορούμε να τροποποιήσουμε ή το λευκό τμήμα του κειμένου που μας υπέβαλε η Επιτροπή τα οποία λευκά τμήματα είναι πολύ πιο δυσχερές να τροποποιηθούν από ό,τι κατάλαβα. Εξεφράστησαν από κάποιες πολιτικές ομάδες κάποιες ε, επιφυλάξεις για το ότι δεν είναι καθόλου αμεληταίος ο αριθμός τροπολογιών που υποβλήθηκαν για το λευκό τμήμα του κειμένου από διάφορους συναδέλφους, δεδομένου του ότι με βάση την ε, διοργανική συμφωνία που υπάρχουν για τις διαδικασίες αναδημιουργίας, αναδιατύπωσης του κειμένου, recast, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για τον τρόπο τροποποίησης. Δύο-τρεις ε, λοιπόν, για να καταστεί ε, σαφέστερη η κατάσταση για τους συναδέλφους. Όντως υποβλήθηκαν αρκετές τροπολογίες για τα λευκά τμήματα, ορισμένες ε, υποστηρίζονται από πολύ ευρείες ε, πλειοψηφίες, ε, δεχομένως και ε, από, το σύνολο των πολιτικών μας ομάδων και σεβαστήκαμε τις φάσεις που προβλέπουν οι διοργανικές συμφωνίες κάθε φορά και το Συμβούλιο και η Κομισιόν ενημερώθηκαν από την Προεδρία της Επιτροπής μας για το ότι θέλουμε να τροπολογήσουμε τα λεγόμενα λευκά τμήματα και αυτή η ενημέρωση επίσης υπήρξε και στην ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπή για όλες τις πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν στην ε, επιτροπή μας. Έγιναν επίσης δύο συνεδριάσεις των σκιωδών, όπου έγινε πολύ ανοιχτή και ευρία ανταλλαγή απόψεων και όπου είχα ζητήσει στους σκιώδεις αν έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες, οι παρατηρήσεις για τα λευκά τμήματα και τις τροπολογίες επ' αυτών. Γιατί βεβαίω είπα ότι είναι αρκετές αυτές οι τροπολογίες επί των λευκών που υποβλήθηκαν από ένα μόνο συνάδελφο και έχω συνέστηση ότι αυτές οι τροπολογίες δεν μοιάζει να την χάνουν ευρεία συνενέσεως. Και ζήτησα κάποιες από αυτές τις τροπολογίες επί των λευκών να ε, αποσυρθούν. Ορισμένες αποσύρθηκαν, αλλά όχι όλες. Διευκρινίζω λοιπόν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Υπήρξε ευρεία δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και για αυτό το λεπτό θέμα των λευκών τροπολογιών που δεν μοιάζει όπως είπα να την χάνουν ευρεία συνενέσως Οπότε τώρα πρέπει να περάσουμε στην ψήφιση. Αλλά με απόλυτα σαφή και διαφανή τρόπο σεβαστήκαμε όλες τις φάσεις της διαδικασίας που προβλέπει η Διοργανική Συμφωνία και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ για αυτή την ε, σαφή εξήγηση. Ξέρω πως είναι περίπλοκο το θέμα. Ευχαριστώ και για τον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκατε. Σημαντική έκθεση τώρα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ξέρω ότι έχουν γίνει ευρείε συζητήσει με την και το Συμβούλιο, οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα προχωρήσει το θέμα αυτό αρχέ του 2013. Ευχαριστώ. Για να ενημερώσω ε, τους συναδέλφους η ψηφοφορία είναι κάπως διαφορετική. Ε, έχει προτείνει η συγκήτρια από κοινού ε, ψήφιση ορισμένων τροπολογιών. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα αρχίσουμε με την αποκοινού ψηφοφορία για τις τροπολογίες που αφορούν την προσωρινή εναπόθεση. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν έχουμε ένα σωρό τροπολογίες για τις οποίες δεν ψηφίζουμε. Ε, έχουμε την τροπολογία 6 της ίντα, νομίζω ότι θα αρχίσουμε την ψηφοφορία σχετικά με την ΙΝΤΑ 6. Ε, έχουμε επιπλέον ψήφους, εγώ δεν θα ψηφίσω. Απορρίπτεται. Έχουμε την ΙΝΤΑ 7 και την τροπολογία 44, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. 45. Όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει διότι ε, ε εγκρίναμε την τροπολογία 1. Δηλαδή, η 45 καταπίπτει νομίζω. Η τροπολογία ανακαλύπτει αυτήν την τροπολογία. Ούτως ή άλλως είναι εύκολη η τροπολογία. Έχουμε την τροπολογία 46, η οποία καταπίπτει και η 47. τώρα περνάμε στην τροπολογία 2, υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 49, υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. 3, υπέρ, καταπίπτει και η 50, 51 καταπίπτουν. 52, συμβατή 52 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, υπέρ, υπέρ, παρακαλώ, κατά, Όχι, όχι. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα από κοινού ψήφιση της τροπολογίας 7 και 55 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 καταπίπτει και τώρα περνάμε στην ίντα 8 υπέρ. Υπέρ, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ίντα 9 καταπίπτει επίσης και η 55. Τροπολογία, όχι, όχι, 55 ήδη περιλήφθηκε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Εντάξει. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μια χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 14 με μια προφορική τροπολογία που θα εξετάσουμε ξεχωριστά. Έχουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της 14 χωρίς το σημείο Β, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που έχουμε εδώ Ψηφίζουμε ξεχωριστά για αυτή την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα ήταν με την προφορική τροπολογία. Πολύ καλά. διότι έχουμε δύο τμήματα. Τώρα έχουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 14, το σημείο Β, εδάφιο Β. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 60 αποσύρθηκε, 62 υπέρ, συμβατή με την τροπολογία 14 υπέρ, κατά εγκρίνεται 61 αποσύρθηκε 64 καταπίπτει α όχι α, επειδή δεν υιοθετήσαμε τη χωριστή ψηφοφορία 64 της κυρίας Ράπτη υπέρ κατά εγκρίνεται 63 65-66 αποσύρονται και 67. Περνάμε στην 68 ε, της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 69 υπέρ κατά εγκρίνεται 70 υπέρ κατά εγκρίνεται 71 υπέρ κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά εγκρίνεται 73 υπέρ κατά εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά εγκρίνεται. Α, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Έχουμε λοιπόν τη 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. Είναι τα 10 υπέρ υπέρ, υπέρ για να δω θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ίντα 10. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, διαγράφεται το άρθρο και τη 75 καταπίπτει, 76 του κυρίου Σβάμπ και την εισηγήτρια υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε με τρεις ψήφους περισσότερους, περισσότερες, 77 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 78 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 17 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται 79 υπέρ, Θα ελέγξουμε και πάλι για την 79, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 80 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 υπέρ, 15 κατά. 81 και 82 ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ κατά. Δεν ήταν σαφή τα πράγματα. Πρέπει να ελέγξουμε νομίζω για 81 και 82 μαζί. Πέρα της ψηφοφορίας. Καλά έκανα και ήλεγξα 18 υπέρ, 17 κατά. 19 κατά πίπτη, 83 αποσύρεται, 84 τροπολογία 20 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Είναι τα 11 υπέρ κατά Οι φιλελεύθεροι ήταν υπέρ, εγκρίνου, ε, ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ο, απορρίπτεται γιατί έχουμε τη μία αποχή. 21 υπέρ. Ας ελέγξουμε και πάλι. Κάποιος έχει κάρτα και δεν ψηφίζει. 20 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται 85 του κυρίου Σμίτ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 86 καταπίπτει και 87 καταπίπτει. Περνάμε στην 88. ...89 επίσης. Υπάρχει μια σύνδεση, μια σχέση. Καταπίπτει επίσης, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα τροπολογιών που καταπίπτουν. 90, 90 καταπίπτει ή όχι. Ε, εγκρίναμε την τροπολογία 20. Ας ε, ψηφίσουμε για την 89, για να βεβαιωθούμε υπέρ. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό έλεγχο. 89. Πέρα στι ψηφοφορία 34 ψήφισαν καταπίπτει. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 90 καταπίπτει, 91 καταπίπτει, τώρα περνάμε στην 22 22 ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. τα 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 92 υπέρ, ας επαληθεύσουμε για την 92. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 υπέρ, 16 κατά, 93 υπέρ, κατά, εγκρίνεται συμβιβαστική α της εισηγήτριας υπέρ, υπέρ της συμβιβαστικής τροπολογίας α εγκρίνεται κατά εγκρίνεται. 94 του κυρίου Σφάμπ υπέρ 98 98, 98 φιλελεύθεροι μπορείτε να με βοηθήσετε η πράσινοι υπέρ κατά εγκρίνεται 99 κατά πίπτη 100 υπέρ κατά πράσινη γκουε, αποχές, εγκρίνεται, ε, με συγχωρείτε, απορρίπτεται, 101 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 102 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 103 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 106 αποσύρθηκε, είναι τα 13 υπέρ, κατά, 107 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 113 καταπίπτει, 114 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 115 υπέρ κατά εγκρίνεται 116 υπέρ κατά εγκρίνεται 117 υπέρ κατά εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ, κατά, ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, 119. Πέρα της ψηφοφορίας, 21 υπέρ, 12 κατά, 120 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 121 αποσύρθηκε, 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 122 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 123 κάνει, είναι μέρος της από κοινού ψήφισης, 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 26 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 124 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 125 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 126 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 127 αποσύρθηκε, 128 και 129 έχουν ήδη ψηφιστεί. Έχουμε μέχρι την 27 του εισηγητή που έχουν ψηφιστεί, 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 139 υπέρ κατά εγκρίνεται 140 υπέρ κατά εγκρίνεται 141 υπέρ κατά εγκρίνεται 142 υπέρ κατά εγκρίνεται 143 υπέρ κατά εγκρίνεται 144 καταπίπτει 28, 147, ταυτόσημες υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 145 και 146 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 148 και 149 και 150 μαζί, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 151 και 152 αποσύρονται 154 υπέρ κατά απορρίπτεται 156 υπέρ κατά εγκρίνεται 155 καταπίπτει 157 υπέρ κατά απορρίπτεται 158 μια διαγραφή υπέρ κατά εγκρίνεται 159 υπέρ κατά εγκρίνεται 160 υπέρ κατά εγκρίνεται 161 υπέρ κατά εγκρίνεται 31 συμβατή υπέρ κατά εγκρίνεται 162 καταπίπτει 163 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, δεχτεί από όλους. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 166 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ, κατά, εγκρίνεται 172 υπέρ κατά απορρίπτεται 173 υπέρ κατά απορρίπτεται 174 υπέρ κατά απορρίπτεται 175 και 176 κίνητα 15 ως είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 καταπίπτει, 179 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 180 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 100 181, 82, 83, 84 όλες μαζί. 33 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. 186 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 187 αποσύρεται. Είμαστε στην 188 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 189 και 190 αποσύρθηκαν. 191 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 35 και οι 16 καταπίπτουν 36 και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 unblock 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές, ε, απορρίπτεται. Η 203 αποσύρθηκε, 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 205 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 37 του εισηγητή, της εισηγητρίας υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 καταπίπτει. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 και 211 αποσύρονται. 38 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τεχνική τροπολογία, την οποία δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 214-215 ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 5. Καταπίπτει. Αυτά λοιπόν. Τελική ψηφοφορία. Συγγνώμη, κάνουμε ένα μικρό έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι δεν μας έχει ξεφύγει κάτι. 17. Ε, να ψηφίσουμε στην τελευταία, για την τελευταία ούτως ή άλλως. Όπως είπα, ελέγχουμε. Α, εντάξει. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Άλλος θα ψηφίσει. 35. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία, δύο αποχές. Μπράβο στην εισηγήτρια. Κυρία Λεγκρίπ, η κυρία Λεγκρίπ και οι σκιώδεις εισηγητές θα συναντηθούν για να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας με το Συμβούλιο και θα επανέλθουν για να μας πούν τι αποφάσεις. Αν έχετε να πείτε κάτι τώρα εδώ στο τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελε απλά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκβαση αυτής της ψηφοφορίας, γιατί νομίζω ότι πραγματικά έχουμε δρομολογήσει μια πολύ θετική διαδικασία ε, και τώρα θα ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα δύο όργανα. Έχουμε λοιπόν ανοίξει το δρόμο για την εμβάθυνση και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Μια προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ για τη λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς. Ε, στον τριμερή διάλογο θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί το λεπτό ζήτημα της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών οργάνων. Πρόκειται για ένα πολιτικό πολύ σημαντικό θέμα ε, και πραγματικά βρισκόμαστε σε πολύ ενδιαφέρουσα θέση από διαπραγματευτική άποψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν δύσκολη η δουλειά σας, πολύ περίπλοκο το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και του σκιώδεις εισηγητές. Ωραία. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ε, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Αντρέας Σβάμπ δεν είναι εδώ. Κυρία Σάνσφερ, θα μας πείτε... Κυρία Σάνσφερ, μήπως θέλετε να πείτε κάτι πριν από την τελική ψηφοφορία. Όχι, θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε κατευθείαν στη γνωμοδότηση. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολο... Συμβιβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, του Κοφεράτη. Τροπολογία 7, χωριστή ψηφοφορία, την οποία ζήτησε το Λαϊκό Κόμμα. Πρώτο τμήμα, χωρίς το κείμενο, σύστημα συλλογικής, ε, συλλογικής προσφυγής, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ. 15 κατά. Η κυρία Βενιόζη είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα επιφωνήματά της. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 10 του κυρίου Ντεγιόγκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. 12. Με μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, του εισηγητή, με την οποία συμφωνούν όλοι νομίζω. Λοιπόν, μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται χωρίς αμφιβολία. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δε... τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αυτή απορρίπτεται 21 υπέρ κατά και αυτή απορρίπτεται 22 υπέρ κατά Αποχές αυτή εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν θα περάσουμε στην ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Πέρας της ψηφοφορίας, 32 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Ο κύριος Ντογιόγκα μου ζήτησε να πω λίγα λόγια. Μήπως η κυρία Χάντσλικ όμως έχει να πει κάτι. Έχετε κάποιο μήνυμα για τον εισηγητή. Απλώς να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας. Εντάξει, ο κύριος Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ να έχει ψηφίσει η Γκουε και να απόσχει στην έκθεση για τον ανταγωνισμό. Αλλά τέλος πάντων χαίρομαι πάρα πολύ που ψήφισαν υπέρ, γιατί ο κύριος Σβέμπ επέδειξε εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας και πραγματικά δέχτηκε και υποστήριξε πολλά θέματα. Πολλές φορές υπάρχει μια έκκληση για απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς σε ομοσπονδιακό επίπεδο ε, και Θέλω να διασαφηνίσω ότι δεν ψήφισα κατά λάθο υπέρ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το υπόλοιπο της έκθεσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Προτείνω να διακόψουμε για λίγο έτσι ώστε να φύγει ο κόσμος και να αρχίσουμε να συζητούμε την γνωμοδότηση του κυρίου Ραμών Όσοι περιμένατε ότι θα, θα ψηφίζατε για την απόσπαση των εργαζομένων, μάθετε ότι έχει αναβληθεί η σχετική συζήτηση. Okay. Merry Christmas and Happy Same to you. Very nice. Thank you for working with us today. Thank you. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas.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 Uh, um, Οπότε, συνάδελφοι, το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, πριν αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Λοιπόν, για να δούμε πολιτικέ ομάδε. Να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών μόλι τελειώσουμε τη ζήτηση αυτού του θέματο. Που δεν νομίζω να είναι πολύ μετά τι 4.30. Δεν νομίζω ότι θα χάσουν πολύ χρόνο. Κυρία Χάνσλεγκ εντάξει. Κυρία Γκέπαρντ, Επίσης συμφωνεί και ο κύριος Μπίλαν. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θέλετε να χάσουμε το χρόνο μας. Όχι, να τον αξιοποιήσουμε σκοπίμως. Αλλά φυσικά δεν πιέζω κανέναν. Δεν πιέζω τον εισηγητή μας. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε αυτά που θα μας πει. Για αυτή τη σημαντική γνωμοδότηση για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες είχαμε δώσει μια σημαντική γνωμοδότηση για την αρχική νομοθεσία που νομίζω ότι επηρέασε τη διατύπωση της πρότασης. Και ξέρω ότι και η κυρία Μακλάχιν έχει εργαστεί πολύ για την πρώτη πρόταση. Με χαρά θα ακούσουμε τη συμβολή της. Υποβλήθηκαν 21 τροπολογίες, θα θέλαμε τη γνώμη σας επί των τροπολογιών και η κυρία Γκάλα έχει μεγάλη πείρα πρώτερη. Ο κύριος Άγκστρομ δεν είναι παρόν, θα έρθει. Η κυρία είναι εδώ, ο κύριος Ντεγιόν δεν είναι πια εδώ. Νομίζω ότι έχουμε μια επίλεκτη ομάδα ε, αφοσιωμένο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Σμιτ. Και όποιος θέλει να συμβάλλει φυσικά μπορεί. Α, μάλιστα. Α, με χαρά ακούμε ότι ενδιαφέρεται και εκείνος. Ο κύριος Σμιτ είναι ασκή και όδους. Ο κύριος Γκαρθές Ραμών. Ευχαριστώ πολύ. Η γνωμοδότησή μου αφορά την εφαρμογή της οδηγίας που σίγουρα είναι πολύ σημαντική για την αγορά οπτικοακουστικών μέσων 10-13. Η γνωμοδότηση που εκπώνησα προσπαθεί να τονίσει τα σημεία που θεωρώ ότι είναι κεντρικά, βασικά, από πλευράς εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και ελπίζω η γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Πολιτισμού που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Έχω τονίσει ορισμένα σημεία. Νομίζω ότι γνωρίζετε ήδη, δεν θα επιμείνω. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Θα επιχειρήσω λοιπόν, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή συνένεση επί των τροπολογιών, να σας εξηγήσω γιατί έχω τα εξής βασικά σημεία. Πρώτον, τονίζω τους κινδύνους συγκέντρωσης και απώλειας ε, διαφορετικών απόψεων, έκφρασης διαφορετικών απόψεων για αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό θα ήταν σοβαρό πρόβλημα για την εσωτερική μας αγορά και τονίζω ότι πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των στόχων της οδηγίας και της ελευθερίας διανομής και πρόσβασης στο περιεχόμενο. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι πολίτες ιδιαίτερος. Τονίζω, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δωρεάν. Επίσης εμένω στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης και την πολιτισμική πολυμορφία για τη δυνατότητα παραγωγής έργων τέχνης, γιατί πιστεύω ότι είναι έφυτο στοιχείο της ελευθερίας έκφρασης αυτό. Και επιμένω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την παραγωγή ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γιατί έχει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στο μέλλον. Μέσω λοιπόν ορισμένων ε, μέτρων πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην εξαφανιστεί στην παγκοσμιοποιημένη αγορά η ευρωπαϊκή παραγωγή. Επίσης πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις ε, διαφημίσεις, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Διότι εμένουν ιδιαίτερα στον εμπορικό χαρακτήρα τα οπτικοακουστικά μέσα. Και μετά υπάρχουν μερικά πιο τεχνικά θέματα. Η σχετική ασάφεια της λέξης πλατφόρμα που αναφέρει επανειλημμένη οδηγία πρέπει να διευκρινίσουμε και τα δικαιώματα χρήσης και κατανάλωσης των προϊόντων στον τομέα αυτό ούτω ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση, πλήρη και ισότιμη. Και κάτι που αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη σε αυτό το τομέα είναι η λεγόμενη διανομή over the top. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές τηλεοράσεις και τους φορείς διαδικτύου πρέπει να διευκρινιστούν. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της ε, γνωμοδότησης που υποβάλλω στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις και να συζητήσουμε για τις τροπολογίες. Κυρία Κάλεβο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω εκφράζοντας τη λύπη μου για το χρονοδιάγραμμα το οποίο ήταν αυτού του φακέλου το χρονοδιάγραμμα διότι για αυτή τη γνωμοδότηση δεν είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δεν είχαμε παρουσίαση της γνωμοδότησης από τον εισηγητή και είχαμε μόνο μια μισή μέρα για την κατάθεση των τροπολογιών. Συνεπώς, λυπούμε, εκφράζω τη λύπη μου, το χρονοδιάγραμμα αυτό, ε, το ότι μας εμπόδισε να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ των εισηγητών. Όπως το είπε ο εισήγητης, αυτή η οδηγία αποτελεί την σπονδυλική στήλη της ρύθμισης της Ένωσης των τομέα ε, των οπτικοακουστικών μέσων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή η οδηγία διατυπώθηκε με τρόπο ώστε να είναι ευστοχή, κέρια, παρά τις ε, τεχνολογικές καινοτομίες εφόσον βασίζεται στην αρχή της ουδετερότητας της τεχνολογικής το κείμενο. Αυτό το ξέρουμε είναι καρπός μακρών και εργοδών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συμβιβασμοί στους οποίους καταλήξαμε είναι ισορροπημένοι και εξυπηρετούν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρηματιών. Η εφαρμογή της οδηγίας έχει αντίκτυπο θετικό πάνω στην ανάπτυξη της αγοράς των οπτικοακουστικών μέσων. Όσον αφορά στις τροπολογίες που κατέθεσα με τους συναδέλφους μου, θα ήθελα ε, να κάνω μερικά σύντομα σχόλια. Πρώτον, μερικές διατάξεις δεν αντιστοιχούν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Συνεπώς κατέθεσα τροπολογίες διαγραφής για τα τρία σημεία που δεν ήταν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, της ΙΜΚΟ. Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΙΜΚΟ, θέλησα πρώτα απ' όλα να τονίσω ε, την συμμόρφωση προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, την αναγκαιότητα της συμμόρφωσης από τα κράτη-μέλη κυρίως όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και την αρχή ε, της χώρας προέλευσης. Δεύτερον, λόγω των νέων μορφών εμπορικής επικοινωνίας που αναφύονται, σκοπεύω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει το 2013 την ερμηνευτική ανακοίνωσή της σχετικά με την διαφήμιση στην τηλεόραση και τρίτον να ενθαρρύνομαι την προσφυγή στο καθεστώς της συρρύθμισης και της αυτορύθμισης που εισάγεται στην οδηγία και που ήδη τα καθεστώτα αυτά, τα συστήματα αυτά έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους, όπως είναι και η ιδεοντολογική κώδικαση ή ή αμερικανική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προσοχή σας. Ναι, σημειώσαμε τα σημεία σας, τις παρατηρήσεις σας. Ε, βεβαίως, ε, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, βεβαίως ε, η απόφαση λήφθηκε αργά σχετικά με την ψήφιση και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Λυπούμε, είναι βεβαίως ε, μια... Είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα την έχουμε τώρα. Ελπίζουμε ε, να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από αυτήν. Ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο Γιούρκεν Κράουτμαν είναι ε, σκιώδης εισηγητής και τον αντικαθιστώ πάντως. Θα διαβάσω μερικές από τις σημειώσεις του ε, σχετικά με την οδηγία η οποία εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη παρόλο που φαίνεται ότι κάπου παραμένουν ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την πλήρη μεταφορά. Η έκθεση εφαρμογής της Κομισιόν δείχνει ότι οι στόχοι της οδηγίας καταρχήν έχουν ικανοποιηθεί η ε, ε, απαγόρευση της ε, προδικαστικής διαφήμισης. Ίσως πρέπει η ερμηνεία, η ανακοίνωση ερμηνευτική να ενημερωθεί από την Κομισιόν. Ωστόσο, όπως τονίζει η Κομισιόν, υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την διαφήμιση, την τηλεοπτική και το όριο των 12 λεπτών ανά ώρα. Η έκθεση αποδεικνύει ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ο κανόνας αυτός παραβιάζεται συστηματικά. Τώρα ο, ο κύριος Κρόσμαν μας λέει ότι μόνο οκτώ κράτη-μέλη έχουν παρακολουθηθεί και δεν ξέρουμε σε πόσα από τα κράτη-μέλη υπήρξαν παραβιάσεις του κανόνα αυτού. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Κομισιό πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα στην πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση εφαρμογής και υλοποίησης είναι ασαφής ως προς το τομέα αυτό. Μια προσωπική παρατήρηση ως προς την απαγόρευση για τα παιδιά ε, και για το ενόπνευμα. Στην χώρα μου υπάρχει μια απαγόρευση. Παρόλο που είμαι φιλελεύθερος, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την απαγόρευση στις διαφημίσεις κυρίως για το ε, ενόπνευμα και για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Αυτή ήταν μια προσωπική παρατήρηση δεν ήταν του κυρίου Κρόιτσμαν, αλλά όπως ξέρετε οι φιλελεύθεροι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις. Τέλος και ίσως αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει ε, την, ε, το πόσο κατάλληλο είναι το πλαίσιο ε, σχετικά με την σύγκληση της κλασικής τηλεόρασης και των διαδικτυακών μέσων θα πρέπει να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις ε, και να δούμε ποιες είναι οι συνήθειες τηλεθέασης των καταναλωτών. Δεν ξέρω αν η οδηγία πρέπει να ε, επανεξεταστεί, αλλά να αναλυθεί η καταλληλότητα των αντιλήψεων και των ορισμών. Γενικό στόχος θα πρέπει να είναι να έχουμε μια ουδέτερα τεχνολογική προσέγγιση, ίσους όρους ε, σχετικά με τις διάφορες συνθήκες για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά των μέσων ενημέρωσης και ε, κλείνω με τις παρατηρήσεις του κυρίου Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε, θέλετε να λάβετε τον λόγο. Κυρία Ρούλε, όχι. Η κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, συζητώντας για το θέμα αυτό. Αυτό που με απασχολεί είναι η καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας και θα ήθελα να κάνω έκκληση στις χώρες μέλη να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν αν δεν το έχουν κάνει. Συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες αυτές να είναι προσπελάσιμες και να υπάρχει μια ελεύθερη πλατφόρμα τηλεοπτική. Δεν μπορώ να υποστηρίξω οι υπηρεσίες αυτές να είναι ελεύθερες δωρεάν, διότι δεν μπορεί να το ζητήσει κανείς από τους οργανισμούς τους ραδιοτηλεοπτικούς και διότι πρέπει να υπάρχουν διάφορα μοντέλα διοδότησης και σύνδρομων. Ε, η κυρία Γκάλαγκερ και ο κύριος Κρόιτσμαν έχουν καταθέσει τροπολογία για να διαγραφεί αυτό το, αυτό το θέμα της δωρεάν παροχής. Ε, δεν ξέρω, ε, ανεξάρτητοι παραγωγές 10-20% προτείνονται στην γνωμοδότηση. Έχω καταθέσει μια τροπολογία που ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν το ελάχιστο όριο όταν αυτό είναι δυνατόν. Για το άρθρο 5 Πιστεύω επίσης ότι οι διευθετήσεις ε, για την, ε, τις διαφημίσεις στα προγράμματα των παιδιών θα πρέπει να επιτυγχάνουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιοτική παροχή και στην προστασία των καταναλωτών. Στην χώρα μου ε, βεβαίως αυτό το θέμα έχει συνέπειες χρηματικές. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν το διαγράψουμε αυτό. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω τα σχόλια της κυρίας Γκάλγκερ για το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και ε, ε, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Μας δώσαν διάφορες ερμηνείες για να εργαστούμε αποτελεσματικά ως ευρωβουλευτές και να μπορούμε να δουλέψουμε καλά. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά, να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Δεν μπορούσαμε ούτε καν να τις καταθέσουμε με το κανονικό σύστημα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό να έχουμε τέτοια πίεση χρονική. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Το ε, θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι το οποίο να είναι έγκυρο, να είναι κατάλληλο για τις χώρες μας. Προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση για το θέμα. Θέλει να λάβει το λόγο κανείς άλλος. Ο κύριος Μπούλουινγκ από την Επιτροπή, από την DG Connect, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε να σχολιάσετε τις τροπολογίες και κάποιες ε, ερωτήσεις και σχόλια για την ε, μεταφορά στο εθνικό εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας. Ευχαριστώ. Θα κάνω κάποια σχετικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Είδαμε το σχέδιο γνωμοδότησης, οι υπηρεσίες της Κομισιόν ε, το εξετάζουν. Ας ξεκινήσω με συγκεκριμένα στοιχεία. Την ιδέα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δωρεάν παροχή τηλεοπτικών, τη οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυμορφία επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου και δεν θεωρούμε ότι είναι καλό να επιβάλλουμε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό ε, μοντέλο. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες υπό την έννοια της οδηγίας συμπεριλαμβάνουν τα συνδρομητικές ε, ε, υπηρεσίες, υπηρεσίες όπως τα iTunes και άλλα θα ήταν πάρα πολύ να επιβάλλουμε να διατίθενται αυτά δωρεάν. Επίσης, ε, η αδυναμία του όρου πλατφόρμα είναι ένα καινούριο θέμα, ένας καινούριος όρος. Ε, υπάρχει η σύγκληση μεταξύ των ε, οργανισμών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και των ηλεκτρονικών μέσων. Πρόκειται να υιοθετηθεί μια πράσινη βίβλος στις αρχές του επόμενου έτους ε, που θα πραγματεύεται αυτά τα θέματα. Η οδηγία οπτικοακουστικών μέσων κάνει λόγο για αυτή την τεχνολογική ουδετερότητα και δεν ασχολείται με τις συσκευές ή τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την παροχή του περιεχομένου. Αυτά ήταν τα τρία γενικότερα σχόλια που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επομένως, επανέρχομαι στον εισηγητή. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο... Α, παρακαλώ. Συγγνώμη, ξέχασα να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας, του κυρίου Σμιτ για τη διαφήμιση. Ε, το είχα γράψει σε, άλλο, σε άλλη σελίδα, με συγχωρείτε η παρακολούθηση των τηλεοπτικών διαφημίσεων είναι παρακολούθηση που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποκαλύπτει κάποια ίσονος σημασίας προβλήματα σε σχέση με τον κανόνα των 12 λεπτών. Βασικά εκ περιτροπής τέσσερα κράτη-μέλη ελέγχονται για την τήρηση του κανόνα αυτού κάθε έτος και συχνά διαπιστώνουμε την παραβίαση του κανόνα των 12 λεπτών. Ε, μόλις ολοκληρωθεί, ε, όταν ολοκληρώνεται η περίοδος της παρακολούθησης ε, ερχόμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη και έχουμε έναν διάλογο όπου απαιτείται ασκούμε τις διαδικασίες για την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και είχε γίνει αυτό πριν από μερικά χρόνια. Ε, το άλλο θέμα για την, μεταφορά, ε, την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο. Ε, θεωρούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του έτους θα μας έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας όσο αφορά την συμφωνία των των εθνικών μέτρων με την οδηγία. Ε, αποστάλθηκαν επιστολές διευκρινήσεων με 20 κράτη-μέλη. Μάλιστα είχαμε διμερείς επαφές ε, για τη διευκρίνηση διαφόρων θεμάτων και δεσμεύσεων και τις περισσότερες φορές ήταν ικανοποιητική η απάντηση. Και πάλι και εδώ, αν η Κομισιόν θεωρήσει ότι δεν πληρούνται οι δεσμεύσει και ότι δεν έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών η οδηγία με το σωστό τρόπο, τότε θα ε, δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ που καλύψατε όλα αυτά. Έχει κάποιο ε, να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Αν όχι, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή να συνοψίσει. Να επιβεβαιώσουμε και το χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία σας δίνω λοιπόν κύριε Ραμόν τον, λόγο. Oui, merci, le président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τις προθεσμίες που έθεσαν διάφοροι συνάδελφοι. Συμφωνώ απόλυτα. Πρώτος εγώ χρειάστηκε να αντιδράσω σε περιορισμένο χρονικό διάστημα που κατέστησαν δυσχερή την εκπόνηση σωστών αντιδράσεων. Δεν υπήρχε δυνατότητα να συνοηθούμε μεταξύ μας. Γιατί χρειάστηκε να υποβάλουμε τις τροπολογίες. Δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε ούτε πριν ούτε μετά την ε, υποβολή των τροπολογιών. Θα πρέπει να συζητήσουμε γενικότερα το θέμα των προθεσμιών. Θα ήταν καλό να επιμηκυνθούν κάπως. Από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, με πολλές ε, συμφωνώ, θα μπορούσα να συμφωνήσω, γιατί βελτιώνουν και εμπλουτίζουν το κείμενό μου, αλλά και κάποιες άλλες. Αν συζητήσουμε μεταξύ μας, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Για δύο-τρεις όμως θα είναι δύσκολο γιατί δεν συμμερίζομαι την άποψη ορισμένων συναδέλφων, γιατί θεωρώ ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της ΙΜΚΟ. Είναι βεβαίως θέματα που είναι στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς. Αφορούν λοιπόν την οδηγία του 2010. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε πώς ακριβώς τίθενται σωστά, πού θα τεθούν για να τεθούν σωστά τα θέματα αυτά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κοινού και για την προστασία μας από τις εμπορικές πρακτικές καθώς και την πρόσβαση. Καταλήγοντας, θα έλεγα Πρόεδρε, καταλήγοντας λοιπόν λέω, ότι έχουμε κάποιο χρόνο μέχρι την, ε, μέχρι την, μέχρι την ε, ψηφοφορία και ελπίζω να καταλήξουμε. Θα ψηφίσουμε μόλις στις 24 Ιανουαρίου. Οπότε έχουμε μόνο τον Ιανουάριο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε χρόνο. Οπότε ξέρουμε στην ε, άλλη επιτροπή η ψηφοφορία θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου. Αλλά ελπίζω να μπορέσουμε, να είμαστε σε θέση δηλαδή, να ψηφίσουμε στις 24. Ε, περιμένουμε εσείς να τους καθοδηγήσετε και Νομίζω ότι και οι θα είναι σε θέση. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγουν έτσι οι εργασίες μας για σήμερα. Η τελευταία συνεδρίαση μας το 2012. ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εργασίες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτούς που μας παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο. Ακολουθεί η συνάντηση των συντονιστών, η οποία δεν μεταδίδεται δημόσια. Ε, ελπίζουμε ε, να συνεχίσουμε να έχουμε την προσοχή σας το 2013. Εύχομαι σε όλους καλή ξεκούραση, ε, καλές χριστουγεννιάτικες διακοπές, το αξίζετε. Uh, Θα ξεκινήσουμε τη συνάντηση με τους συντονιστές μόλις